on l'ai vu les jours même. Merci. Dear colleagues, it is uh, time... Συνάδελφοι, ώρα να ξεκινήσουμε. Διότι έχουμε πολύ φορτωμένη μισή διάταξη. Item 6 uh, in our agenda. Σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Ενημέρωση για τις οργανικές διαπραγματεύσεις για τον τρίτο διάλογο, τον διάλογο η οδηγία ΝΕΚ που έγινε χτες η συζήτηση το απόγευμα στο τριμερή διάλογο. Συζητήθηκαν διάφορες διατάξεις όπως και υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βάλει εκθέσεις, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, πληροφορίες και κυρώσεις. Και στο δεύτερο τριμερή διάλογο προχώρησαν τα θέματα αφού ε, έγιναν πρόοδοι στο τεχνικό επίπεδο. Στο παράρτημα 2 των δεσμεύσεων για εκπομπέ σε εθνικό επίπεδο, για μείωση των εκπομπών, το Συμβούλιο είπε ότι ερχόταν σε διμερεί επαφέ με τα κράτη-μέλη, ώστε να αναθεωρηθούν τα διάφορα στοιχεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση επεσήμανε προθυμία να συμφωνήσει να μειώσει την τροπολογία του για την πρώτη δέσμευση για μειώσει σε 20% των εκπομπών. Όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους, έγινε 7ο τριμερής διάλογος την 9η Απριλίου. Το εισηγητή ενημέρωσε το Συμβούλιο Διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΜΒΗ και Άγκρη για το θέμα των ελέγχων στον οργανικό τομέα. Η διαπραγματευτική ομάδα συζήτησε διάφορα άρθρα με προϋποθέσεις για επισήμους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες σε διάφορους τομείς. Δόθηκαν διευκρινήσεις όσον αφορά τους συμβιβασμού που προτείναμε το Φεβρουάριο του 2016. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν επικοδομητικά. Παραμένει το θέμα της, εξουσο... της ανάθεσης των εξουσιών. Η συζήτηση συνεχίστηκε με εξέταση των διαφόρων διατάξεων που αφορούν την επιβολή των μέτρων. Ο εόδος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πολύ ε, μεγάλη περίοδο ψηφοφοριών. Παρακαλώ να βάλετε τις κάρτες για τις ψηφοφορίες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα όρια κομπών και εγκρίσεις τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσεως. Για... Η Ελιζαβέτα Γκαρντίνη ε, συμφώνησε ε, με τους άλλους συνομιλητές μετά από πολύ μακρά διαδικασία. Έχουμε τη συμφωνία της πρώτης ανάγνωσης και θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Avete votato tutti. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα. Α, συγχαρητήρια στη συνάδελφο Γκαρντίνη. Και τώρα πάμε στην ψηφοφορία που αφορά το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση πρόοδου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξεκινάμε αμέσως την ψηφοφορία. Πρώτη ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται α, έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 8, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Οι σοσιαλιστές δεν έχουν δύναμη στο χέρι, δεν σηκώνουν πολύ το χέρι. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. εγκρίνεται Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 45 όχι, 46, καταπίπτει 45. 46 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, τροπολογία 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται Εξήντα έξι, τροπολογία εξήντα έξι. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 103. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εκκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Και τώρα πάμε. Ο Πίτερ. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω ε, κάτι για αυτήν την ε, γνωμοδότηση για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τη συνάδελφο και τους Κιώδης. Έχουμε μια καλή βάνη. Ε, ένα λεπτάκι, Πίτερ, γιατί δεν, δεν έχουμε αγγλική μετάφραση. Θα τα πω στα αγγλικά λοιπόν. Ευχαριστώ λοιπόν ε, τους ε, σκιώδεις. Νομίζω ότι έχουμε μια καλή βάση ε, για αυτή την ψηφοφορία. Απλά ήθελα να ανακοινώσω κάτι τεχνικό. Η τροπολογία 39 στην παράγραφο 4 συμφώνησα με την κυρία Γκίζετεγκ ότι θα μπορούσε να γίνει ψηφοφορία πρόσθετη, συμπληρωματική. Θα γίνουν κάποιες ε, διαγραφές δηλαδή, απλά ότι αυτά θα προσθεθούν στην, στην παράγραφο 4 και άρα αυτή η, σύσταση απλά προστίθεται στα όσα ήδη υπάρχουν και έχουμε ελέγξει το θέμα και με τη γραμματεία. Άρα η 39 ε, ε, θα ψηφιστεί ως προσθήκη στην παράγραφο 4. Ευχαριστώ. Thank you. Before the vote, Ευχαριστώ πριν ψηφίσουμε. Θα θυμηθώ το αίτημα του εισηγητή και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα συμφιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την 39 ως εξηγήθηκε από τον συνάδελφο Λίζε σαν προσθήκη στην παράγραφο 4. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμφιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω χέρια από τους σοσιαλιστές. Επαναλαμβάνουμε. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 88 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 103 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 105 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνατε. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 109 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 113 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή, τον κύριο Λίζε. punto 10 all'ordine del giorno. 10 της ημερήσιας διάταξη. Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης. Ξεκινάμε λοιπόν στη συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τροπολογία 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Επαναλαμβάνουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα. Τροπολογία 70. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά άποχες αγαπητοί συνάδελφοι υπάρχει ένα πρόβλημα δεν έχουμε τους σοσιαλιστές στην αίθουσα επαναλαμβάνουμε διότι αν λείπει μια μικρή ομάδα, εντάξει το καταλαβαίνουμε. Αν λείπει μεγάλη ομάδα, παρακαλώ να σηκώσετε το δάχτυο, το χέρι. Να. Υπέρ της 72 παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 84 και την 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 και 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 9. Όχι, καταπίπτει. Την 91 πιετικάνεν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα τη συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 103 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ Το πρώτο τμήμα, ζητώ συγγνώμη, καταπίπτει. Το δεύτερο τμήμα, συμβατό με την τροπολογία 102. Ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 104. Υπέρ, κατά, άποχες, έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι μάλλον απορρίπτεται, αλλά το ελέγξουμε. Ψήφισαν όλοι, πέρας, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 106. Α, πάμε στην 109. Τροπολογία 109 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 110 απεσύρθη, συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αν θέλετε τον έλεγχο, τον κάνουμε λοιπόν. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Γιατί συμβιβαστική 5. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Τώρα, στην 131 πάμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Την 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβαστική 8. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 146 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, εγκρίνεται.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 αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά έλεγχος Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά άποχες έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Εντάξει, αφού θέλετε. Έλεγχος λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Άρα τώρα πάμε στην τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τοπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά θα κάνουμε την τελική ψηφοφορία που ξεκινάει. Avete votato tutti? No, qualcuno non vota. Il voto è chiuso. Approvato. E Congratulazioni λοιπόν. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Possiamo passare al prossimo... Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μας με τις μετεκλογικές αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Ξεκινάμε αμέσως. Συνάδελφε Γκάμπους, είσαστε εισηγητής. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. Ψηφίζουμε λοιπόν σε δύο τμήματα την τροπολογία 17, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 19, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πρέπει λοιπόν τώρα αν θέλετε να κάνουμε έναν έλεγχο γιατί 19 το κάνουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έλεγχος λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Παρακαλώ να ψηφίσετε την τροπολογία 18, διότι η τροπολογία 14 απερίφθη. Συνεπώς, πείτε μου ποιος είναι υπέρ της 18. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 σε δύο τμήματα. πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 25 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στο σημείο 12 all'ordine del giorno. Σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ξεκινάμε. Συμβαστική 1 υπέρ συμβαστικής 1 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 17 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπερ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπερ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική 4. Υπερ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, απορρίπτεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 με προσθήκη στη 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 54 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 55 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 56 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. Τώρα διακόπτουμε για ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Για μία ώρα διακόπτουμε. Και τέταρτο, θα έχουμε την Επίτροπο Μπούλτς στις 5 και τέταρτο. Yeah. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ε, ανταλλαγή απόψεων με την ε, κυρία Βιολέτα Μπούλς, Επίτροπο Αρμόδια για τις ε, Μεταφορές σχετικά με την πιθανότητα παγκόσμια αγορακεντρικού μέτρου ε, για τη μείωση των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα από την αεροπορία. Καλωσορίζω θερμά την κυρία Βιολέτα Μπούλς ε, στην Επιτροπή μας για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Η επόμενη συνάντηση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, ΙΚΑΟ, θα πραγματοποιηθεί στο Μόντρεαλ από 11 έως 13 Μαΐου. Και θα ε, παρευρεθεί και αντιπροσωπεία της Επιτροπής ε, ΕΝΒΗ. Να σας θυμίσω ότι όλα τα θεσμικά πλάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήθελαν να συμπεριληφθεί η αεροπορία στην ε, Συμφωνία του Παρισιού, κάτι το οποίο όμως δεν ήταν δυνατόν στο τέλος. Το θέμα αυτό συζητήθηκε και κατά το Κοινό Συμβούλιο Περιβάλλοντος και Μεταφορών τον Απρίλιο στο Άμστερνταμ. Επιπλέον, επειδή εκπνέει η νομοθεσία Stop the Clock ε, για τις ε, διπυρωτικές πτήσεις, Τα επόμενα βήματα θα εξαρτηθούν από την απόφαση του ε, Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας ε, για ε, το Παγκόσμιο Αγορακεντρικό Μέτρο. Είναι σημαντική αυτή η συμφωνία για ε, την ε, αεροπορία. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε την ε, θέση σας για τις διαπραγματεύσεις και πώς βλέπετε την κατάσταση των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα και μπορούμε ως συνήθως να ξεκινήσουμε από τη δική σας παρουσίαση. Σας δίνουμε 10 λεπτά και κατόπιν θα έχουμε δύο γύρους ερωτήσεων και απαντήσεων. Πρώτα θα ακούσουμε τους ε, συντονιστές των πολιτικών ομάδων ε, και κατόπιν θα ακούσουμε ε, τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίδετε τη δυνατότητα για πρώτη φορά να παρευρεθώ εδώ στην Επιτροπή σας. Ελπίζω ότι θα είναι επικοδομητική η συζήτησή μας, διότι αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις. Οι προκλήσεις είναι σημαντικές, ε, μας δίνουν όμως και την ευκαιρία να κάνουμε κάτι σημαντικό για το μέλλον. Όχι μόνο του πολιτισμού μας, αλλά και του πλανήτη. Ε, η συμβολή της ε, αεροπορίας ε, στην μείωση των εκπομπών είναι σημαντική. Το 2% μερικοί θεωρούν ότι είναι μικρό ποσοστό, αλλά θα είναι σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε σοβαρά με τα στοιχεία αυτά. Χαίρομαι λοιπόν που θα συμμετέχετε κι εσείς στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, συνάντηση υψηλού επίπεδου ε, της το στο Μόντρεαλ τον επόμενο μήνα. Η συνάντηση του Φεβρουαρίου ήταν σημαντική για μένα. Συνάντησα ε, ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις, που διαπραγματεύονται τα έγγραφα τα οποία συζητάμε και έτσι έχουμε καλύτερη κατανόηση του τι ε, μπορούμε και τι θέλουμε να πετύχουμε όλοι μαζί. Πιστεύω λοιπόν ότι και η συνάντηση του Μαΐου θα συμβάλλει εξίσου σημαντικά στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων. Η συμβολή της αεροπορίας στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος είναι ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα το οποίο συζητήσαμε και στο άτυπο Συμβούλιο Μεταφορών και Περιβάλλοντος ε, στο Άμστερνταμ πριν 10 μέρες. Ήταν ε, σημαντικό το ότι συζητήσαμε ακριβώς ε, τα θέματα αυτά. Ελπίζω αυτό να γίνει συνηθισμένη πρακτική και στο μέλλον. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την αλλαγή του κλίματος είναι πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά. Πέρα από τη συζήτηση για το πού οφείλεται η αλλαγή του κλίματος. Ε, το γεγονός είναι ότι το κλίμα αλλάζει. Ε, βλέπουμε ότι λιώνουν οι πάγοι, ότι ε, ανεβαίνει το επίπεδο των θαλασσών. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε την πλήρη έκταση των φαινομένων αυτών, διότι θα επηρεάσουν τη ζωή μας. Συμφωνήσαμε ότι η αεροπορία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη ε, Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, αλλά να βρούμε και λύσεις ώστε να αντισταθμίσουμε τις αντικές συνέπειες ε, της ανάπτυξης. να έχουμε ανάπτυξη με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, αλλά να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί όχι μόνο στην αγορά εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι ο ΙΚΑΟ είναι ο ε, κατάλληλος οργανισμός ε, να κάνει τις διαπραγματεύσεις, ε, διότι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, απαιτείται και παγκόσμια λύση. Δεν θα πρέπει να βασιστούμε μόνο όμως στις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να έχουμε καλύτερη διαχείριση Έχουμε τώρα το εργαλείο Σεζάρι για την αποτελεσματική διαχείριση ε, της κυκλοφορίας, αλλά θα πρέπει επίσης ε, να προσέξουμε τις εξελίξεις ε, όσον αφορά τις τεχνολογίες που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το βλέπουμε και στην αεροπορία. η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι μόνο με νομοθεσία και καλύτερη αποτελεσματικότητα θα μπορέσουμε να πετύχουμε ε, τις αλλαγές που είναι απαραίτητες για να πετύχουμε το στόχο των ε, μηδενικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα αλλά με την ε, σύγχρονη τεχνολογία μπορούμε να το πετύχουμε και γι' αυτό ε, βρίσκω συναρπαστική την είδηση ότι ε, έχουμε το πρώτο υβριδικό αεροπλάνο. Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τον τομέα να ακολουθήσει τις αλλαγές αυτές και να εισάγουμε και τις αλλαγές που σας ανέφερα στους άλλους τομείς σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή των αερομεταφορών από ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ε, παίζουν και τα αεροδρόμια και έχουν κάνει σημαντικά βήματα όσον αφορά τις δραστηριότητες τους. Ε, για παράδειγμα, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που να βασίζεται σε βιώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα από τα κλειδιά για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ε, ανάπτυξη στη φάση αυτή μέχρι να πετύχουμε ε, σημαντικές νέες πρόοδους στην τεχνολογία. Όπως ήδη αναφέρθηκε, δεσμεύομαι προσωπικά να ε, εργαστώ με στόχο μια φιλόδοξη συμφωνία στην συνέλευση του ΙΚΑΟ ε, παρουσιάζοντα τα αποτελέσματα που συμφωνηθήκαν ε, στον ΙΚΑΟ το 2013. Συνεργαζόμαστε στενά με τον Πρόεδρο Άλιου και ε, εταίρους από τρίτες χώρες για να πετύχουμε το σημαντικό αυτό στόχο. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχουμε την πρόταση του Πρόεδρου Αλίου. Ε, υπέβαλε την πρόταση αυτή πέρσι τον Δεκέμβριο και ε, έχει τροποποιηθεί τα, τους τελευταίους μήνες, έχει βελτιωθεί και Παρά όμως ε, τις ε, ισχυρές ε, επικρίσεις από κάποιους ενδιαφερομένους, ο Πρόεδρος κατάφερε να αποτελεί αυτό το μόνο κείμενο διαπραγματεύσεων, κάτι που επικροτούμε. Πρέπει να έχουμε ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο που να αντισταθμίζει τις ε, αρνητικές συνέπειες ε, και νομίζω ότι μπορεί το κείμενο αυτό να αποτελέσει πολύ καλή βάση για τις διαπραγματεύσεις και να βελτιωθεί περαιτέρω. Η πρόταση του Προέδρου ε, πετυχαίνει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε διάφορες πτυχές. Καταρχάς, την μη διάκριση. Λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, διατηρώντας ε, όμως ε, και την περιβαλλοντική ακαιρεότητα. Πιστεύουμε ότι οι αερομεταφορείς θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση στις ίδιες διαδρομές, διότι έτσι μειώνουμε στο ελάχιστο τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ανάμεσα στις δικές μας επιχειρήσεις και αυτές των τρίτων χωρών. Επίσης, ε, θέλουμε σταθεροποίηση των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα ε, από την διεθνή αεροπορία μέχρι το 2020. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω τρία πολύ σημαντικά στοιχεία που ελπίζουμε ότι θα ενισχύσουν την πρότασή μας. Καταρχάς, θέλουμε ε, τα βασικά στοιχεία του αγορακεντρικού μέτρου ε, να ε, μας δώσουν ανάπτυξη με ουδέτερο ζύγιο άνθρακα μέχρι το 2020. Δεύτερον, η πρόταση επιτρέπει περιοδικές αναθεωρήσεις, κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ ισχυρό εργαλείο, διότι έτσι δεν δεσμεύομαι σε μία μοναδική και τελική λύση. Επιτρέπουμε τις ε, αναθεωρήσεις ώστε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε. Δεν ε, θα κλείσουμε δηλαδή μια συμφωνία και δεν θα αλλάξει τίποτα τα επόμενα 20 ή 30 χρόνια. Μας ε, επιτρόπει περιοδική αναθεώρηση, το να βελτιώνουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και επίσης ε, θα πρέπει να βασίζεται ε, σε διατάξεις ε, διαφάνειας, δηλαδή να έχουμε μετρήσεις, αναφορές και επαλήθευση, MRV, και να έχουμε αντισταθμιστικά μέτρα υψηλής ποιότητας, ώστε να έχουμε πραγματική μείωση των εκπομπών καθότι δεν ε, θα συμφωνηθούν όλα τα στοιχεία του αγορακεντρικού μέσου από την ε, συνέλευση. Το σχέδιο ψηφίσματος θα πρέπει να περιλαμβάνει και έναν οδικό χάρτη με τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να οριστικοποιηθούν ε, εγκαίρως, ώστε το αγορακεντρικό μέσο να αρχίσει να λειτουργεί από το 2020 και μετά. Πολύ σημαντικοί παράγοντες και εταίροι ήδη στηρίζουν την πρόταση του Προέδρου αλλά πρέπει να πούμε ανοιχτά ότι δεν συμφωνούν όλοι ακόμα. Απαιτούνται λοιπόν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Τα καλά νέα είναι όμως ότι ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάρει θέση ανοιχτά είναι υπέρ της επίτευξης μιας συμφωνίας. Έχουμε κάνει λοιπόν σημαντικό βήμα από το σημείο που βρισκόμασταν στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Έχουμε λοιπόν τη δέσμευση, θέλουμε να ε, εκμεταλλευτούμε την ε, θετική ενέργεια της Συμφωνίας COP21 και είμαι πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση τελικά. Αλλά θα χρειαστεί σημαντική προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις και γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε ενωμένοι, να παρουσιάσουμε τις θέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ταυτόχρονα να είμαστε ευέλικτοι και να δείξουμε ότι κατανοούμε τις ε, λύσεις που παρουσιάζονται. Ποιες είναι λοιπόν οι προσδοκίες μας από τις διαπραγματεύσεις. Καταρχά, ο στόχος ε, του ΙΚΑΟ είναι να πετύχουμε ανάπτυξη με δεύτερο ισοζύγιο άνθρακα στην αεροπορία από το 2020. Αυτό λοιπόν ε, είναι το βασικό μας κίνητρο. Αρχικά είχαμε πιο φιλόδοξο στόχο, αλλά έχοντας κατά νου τι δύσκολες διαπραγματεύσεις μπροστά μας, ας ε, κάνουμε πρώτα αυτό το πρώτο σημαντικό βήμα. Εάν συμφωνήσουμε ότι έχουμε μία πολύ ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε και εάν έχουμε και τις ε, περιοδικές αναθεωρήσεις χρησιμοποιώντας ε, το μοντέλο που συμφωνήθηκε στο Παρίσι στη Συμφωνία COP21 ε, θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή διαδικασία στη συνέχεια. Πιστεύω λοιπόν ότι το Παγκόσμιο Αγορακεντρικό Μέτρο, το GMBM, αποτελεί εργαλείο για να πετύχουμε το στόχο αυτό με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Εάν υιοθετήσουμε και σας καλώ να με στηρίξετε αυτό. Εάν ε, συμφωνήσουμε ότι ό,τι συμφωνήσουμε τον Οκτώβριο δεν θα είναι το τελικό προϊόν, ε, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ περισσότερη επιτυχία. Η συνέλευση θα πρέπει να υιοθετήσει ένα ψήφισμα το οποίο καθορίζει τις ε, κατευθυντήριες αρχές ε, για ένα μελλοντικό παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι το 2020. Ο ΙΚΑΟ κατόπιν θα πρέπει να αναπτύξει όλα τα επιμέρους στοιχεία και τα εργαλεία εφαρμογής ώστε να λειτουργήσει αυτό το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται σκληρά σε προετοιμασία της συνέλευσης ώστε να είναι όσο γίνεται πιο ε, στεναρά τα υπόλοιπα στοιχεία. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε διεθνείς διαπραγματεύσεις ε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δεν συμμερίζονται τις θέσεις μας ε, και έτσι θα είναι σημαντική πρόκληση το να πετύχουμε όλους τους στόχους μας. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να παραμείνουμε φιλόδοξοι, πρέπει όμως να είμαστε και ευέλικτοι και διατεθειμένοι να πετύχουμε συμβιβασμούς ή κάτι που προτιμώ ακόμα περισσότερο να βρούμε νέες λύσεις που να βασίζονται στις διάφορες ε, ε, απόψεις. Για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί με άλλους ε, σημαντικούς παράγοντες με τρόπο ανοιχτό και αποτελεσματικό. Θα πρέπει να δράξουμε κάθε ευκαιρία για να πείσουμε τους άλλους και να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας σε όσους δεν ε, έχουν πιστεί ακόμα ότι είναι απαραίτητο ένα αγορακεντρικό μέτρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη, στο σύνολό της, ε, δημιουργεί επαφές με διάφορους εταίρους και σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο. Και σας διαβεβαιώ ότι δράτω με κάθε ευκαιρία να παρουσιάσω τις θέσεις αυτές σε εταίρους μας. Ε, χθες, για παράδειγμα, ε, ε, συναντήθηκα με τον Υπουργό Φόξ και συμφωνήσαμε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε να είναι ενωμένοι για να μπορέσουμε να πείσουμε και τους υπολείπους. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είναι ισχυροί εταίροι και ότι θα μπορέσουμε έτσι να ε, συνεχίσουμε επιτυχώς τις διαπραγματεύσεις. Ήδη σας ανέφερα την επίσκεψή μου στο Μοντρεάλ τον Φεβρουάριο, όπου συναντήθηκα με ε, όλους τους πρέσβεις, τους πρέσβεις ε, της Ευρώπης, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από χώρες του υπόλοιπου κόσμου και είχα την αίσθηση ότι όλοι θέλουν να πετύχουν συμφωνία και γι' αυτό είμαι πεπισμένη ότι με ανοιχτό διάλογο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Μία από τις πιο σημαντικές επικείμενες επισκέψεις θα είναι το ταξίδι μου στην Κίνα όπου θα θίξουμε το θέμα απέναντι στους εταίρους και συναδέρφους μας στην Κίνα. Η Κίνα δεν έχει εκφράσει ακόμα σαφώ τη θέση της. Το ίδιο κάνουμε στην περιοχή του Κόλπου, στη Σιγκαπούρη, όπου την οποία επισκεφτήκαμε αρχές της χρονιάς. όπου βλέπουμε ίσως όχι ενθουσιώδη υποστήριξη, αλλά βλέπουμε ότι παίρνουν σοβαρά το θέμα αυτό και ότι θέλουν να πετύχουν πρόοδο. Το ίδιο ισχύει και για την Αιθιοπία όπου είχαμε συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με την Αφρικανική Ένωση. Χαιρόμαστε λοιπόν που και η Αφρική ε, επιθυμεί τη σύναψη συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει επιδείξει ενότητα μέχρι τώρα. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλλει σε καλύτερη λύση. Χαίρομαι όμως που κρατάμε ανοιχτό το διάλογο, ότι συντονίζουμε τις θέσεις μας και είναι σημαντικό η διεθνής κοινότητα να νιώθει ότι ε, ε, ε, ότι διαπραγματεύεται με έναν ισχυρό εταίρο και πιστεύω ότι αυτό θα επηρεάσει θετικά το τελικό αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ ευχαρίστως θα συνεχίσει να ε, σας υποβάλει εκθέσεις ε, σχετικά με την πρόοδο, εφόσον σας ενδιαφέρει. Σας παρακαλώ ενημερώστε με. Ε, αν θέλετε να συναντηθούμε πάλι πριν το φθινόπωρο, πολύ ευχαριστώ, θα ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο αίτημα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα στο τέλος να ξανατονίσω πόσο σημαντικό είναι να είμαστε αποφασισμένοι, να έχουμε μια λογική αντιμετώπιση και να μιλάμε ανοιχτά με όλους τους εταίρους μας, διότι όπως λέει ο πρόεδρος Αλιού και συμφωνώ μαζί του, καμία χώρα δεν θα πρέπει να μείνει πίσω στη διαδικασία αυτή και το πιστεύω αυτό πραγματικά. Εάν θέλουμε να συμβάλλουμε σημαντικά στην ε, απαλλαγή της βιομηχανίας από εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, θα πρέπει να δώσουμε σε όσους δεν είναι έτοιμοι τώρα να συμμετάσχουν πλήρως σε μια μεταβατική περίοδο. Εάν το έχουμε αυτό κατά νου, είμαι πεπισμένη ότι θα πετύχουμε μια συμφωνία πάνω στην οποία θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως με τις πρώτες ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο Πίτερ Λίζε από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την ανταλλαγή απόψεων και για τον ανοιχτό τρόπο με τον οποίο συζητάτε αυτά τα θέματα με το Κοινοβούλιο. Οπότε σας ζητάτε και ε, θα, θα είναι απαραίτητο βεβαίως και στο μέλλον κάτι τέτοιο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταλήξουμε σε μια ιδανική λύση. Είπατε λοιπόν ότι με τα ε, μέλη του επιτελείου σας διαπραγματεύονται εδώ και 10 χρόνια αυτό το θέμα. Ε, ε είχαμε συζητήσει το 2006 την πρώτη πρόταση της Κομισιόν. Ο Ματίας Γκρότε ήταν τότε σκιώδης ε, εισηγητή σε μια έκθεση που συνέτασα εγώ και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να καταλήξουμε σε μια τέτοια συμφωνία. Πρέπει να δούμε τι είναι επιστημονικά εφικτό και απαραίτητο. Το καλό είναι ότι η ένταξη της αεροπορίας στο ETS στην Ευρώπη επετεύχθη η ε, Κίνα, η Ινδία, η ΙΠΑ δεν θέλαν ε, να καταρτιστεί ένα τέτοιο σύστημα παγκόσμια, αλλά στην Ευρώπη το ακολουθούν. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικές σημειώσεις των εκπομπών μέσω του ETS σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντική η συμβολή της αεροπορίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου καταφέραμε να εφαρμόσουμε ε, τον δικό μας κανονισμό. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα πρέπει να μπούμε σε συζητήσεις για το αν θα το καταργήσουμε εμείς. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσουμε το ETS. Το τι θα κάνουμε εκτός Ευρώπης βεβαίως είναι διαφορετικό και πιο ε, δύσκολο ως θέμα γιατί θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον ICAO. Και στόχος μας θα πρέπει να είναι να ε, προωθήσουμε προ τη σωστή κατεύθυνση τον ΙΚΑΟ και όχι να δώσουμε πατήματα σε εκείνου που θέλουν να κάνουν τα αντίθετα με εμάς. Φυσικά, μπορεί κανείς να πει ότι 2% ε, Άλλοι εμπειρογνώμονε ε, μπορούν, να έχουν διαφορετική γνώμη, αλλά βλέποντας και μόνο το διοξίδιο του άνθρακα, είναι εντυπωσιακό πως μεταξύ των 180 κρατών που υπέγραψαν τη Συμφωνία των Παρισίων, μόνο οι 129 και χωρίς μάλιστα την Κίνα και τις ΗΠΑ, 129 χώρες λοιπόν, αφρικανικές, λατινοαμερικάνικες, ασιατικές χώρες, οι εκπομπές από αυτές τις 129 ε, χώρες είναι λιγότερες από ό,τι αυτές που οφείλονται στην διεθνή αεροπορία. Διαρκώς επαναλαμβάνουμε λοιπόν τα επιτεύγματα των Παρισίων και τις 180 χώρες που υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την συμβολή της αεροπορίας, διότι είναι μεγαλύτερη από, ε, ε από ότι η συμβολή 129 χωρών όπως είπα. Και αυτή τη στιγμή ο ΙΚΑΟ μιλάει για ανάπτυξη με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Δυστυχώς η, η παρότι δέχτηκε ε, μια σειρά από ζητήματα, ο ΙΚΑΟ το μόνο που δέχτηκε ήταν οι αντισταθμίσεις και είναι βεβαίως σημαντικό να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά δεν θα συμβάλλει ο κάθε αερομεταφορέας στην ανάπτυξη με ιδιαίτερο ισοζύγιο άνθρακα. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία λέει ότι θα αφήσουμε κάποιο περιθώριο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εγώ θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι ναι πρέπει να δημιουργήσουμε, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, αλλά να μην έχουμε αυταπάτες. Ο ΙΚΑΟ δεν είναι η οργάνωση που θα λύσει το πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχει διάταξη αναθεώρησης και να προχωρήσουμε σε διμερές υπόπεδο με διάφορους εταίρους, ε, για παράδειγμα και με τον, ε, η επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία και θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε το δικό μας σύστημα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γκρότη για τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπούλς που μας προσφέρετε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας σήμερα. Το περιγράψατε. Ε, ότι ε, στόχος είναι μια ανάπτυξη με ιδιαίτερο ίδιο άνθρακα. Ε, εγώ σκέφτομαι το εξής. Πώς θα το πούμε αυτό σε άλλους ε, κλάδους και σε άλλες βιομηχανίες. Ε, συζητούμε ε, τις μειώσεις των εκπομπών. Και μάλιστα είμαστε και πολύ αυστηροί. Αν μας πούν οι άλλοι κλάδοι λοιπόν ότι ε, θέλουμε να αναπτυχθούμε και εμείς με ουδέτερο ισοζυγείο άνθρακα, δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους ε, πείσουμε για, για κάτι τέτοιο. Τι λύσεις θα μπορούσατε να, ε, να, να τους προτείνουμε. Πώ πιστεύετε ότι μπορεί να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στον ΙΚΑΟ ε, που να είναι βιώσιμη και που να μπορεί να πείσει και τους άλλους κλάδους. Ο Ιεν Ντάγκαν θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες αν για άλλη μια φορά θεσπιστούν τρομερές εξαιρέσεις για την αεροπορία. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν δεν ακολουθήσουμε ε, ευρωπαϊκό, ε, την ευρωπαϊκή οδό, τότε θα, θα, θα βάλουμε άλλο ένα καρφί στη σαρκοφάγο του ευρωπαϊκού οράματος. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ώστε να ενισχύσουμε το δικό μας ε, ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών και να δείξουμε και στους εταίρους μας ότι ένα τέτοιο σύστημα για μας είναι απαραίτητο στοιχείο μιας διεθνούς συμφωνίας και δεν τη συζητάμε καν. Ευχαριστώ πολύ για το ECR η κυρία Γκέρλιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όταν θεσπίστηκε ο μηχανισμός αναστολής. Ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και από το να ζητούμε απλά το πώς θέλουμε εμείς να είναι αυτό το σύστημα και τι μορφή θα πρέπει να έχει αυτή η συμφωνία ε, δεν θα μας βοηθήσει ούτε θα μας ε, πάει πολύ μπροστά ε, Χαίρομαι που είπατε ότι ένα τέτοιο παγκόσμιο μηχανισμό μπορεί να μην είναι ιδανικό ή τέλειο από την αρχή, αλλά ότι είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα και ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα των αναθεωρήσεων. Και νομίζω ότι ε, βρισκόμαστε σε μία από αυτές τις περιπτώσεις όπου το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Τι νόημα θα είχε ένας παγκόσμιος μηχανισμός αν διατηρήσουμε και έναν περιφερειακό μηχανισμό. Αυτό θα είναι πάρα πολύ, δύσκολο ως θέμα και για την Κομισιόν και για το Κοινοβούλιο. Και αυτό δεν αφορά μόνο το μετριασμό της κλιματικής αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουμε τα δυνατά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συμφωνήσει ότι η φιλοδοξία για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από το 2020 και έπειτα δεν είναι και ιδιαίτερα φιλόδοξη, δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλή. Αλλά αν πάρουμε υπόψη μας την αφετηρία από την οποία ξεκινήσαμε, δεν είναι και αμεληταία αυτή η διαδικασία. Πιστεύετε εσείς, όταν ήμασταν στο, ε, στο Παρίσι και συζητήσαμε την κλιματική αλλαγή, είχαμε ε, καταλήξει και στο θέμα της ε, κοινή ευθύνης της κοινή περιβαλλοντολογικής ευθύνης και με βάση αυτήν καταλήξαμε και σε μια στρατηγική του ΟΗΕ. Αν αυτό το θέμα ε, επαναληφθεί και ενσωματωθεί και σε αυτό το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο, ακόμη και αν λάβει κάποιο, κάποιο, κάποιο, άλλο όνομα, ειδικέ περιστάσεις ή οτιδήποτε, θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μια λύση ιδανική. Θα χρειαστούν διαπραγματεύσεις και αλλαγές. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι τι θα γίνει με τα μέτρα μετριασμού για τις ενδοευρωπαϊκές Έχετε κατά νου κάποιους άλλους ε, μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Έχουν εξφραστεί διάφορες απόψεις. Αλλά ε, έχετε υπόψη σας κάποιες άλλες λύσεις που δεν έχουν σχέση με αγορακεντρικά μέτρα ή με το ETS. Θα ήθελα τη γνώμη σας από αυτό. το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε. Ευχαριστώ για τα αρχικά σας σχόλια. Είπε η Τζούλη ότι το τέλειος είναι εχθρός του καλού. Αλλά ε, η έλλειψη φιλοδοξίας ίσως να είναι η άρνηση ενός λαμπρού μέλλοντος. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Θα μπορούσα να επαναλάβω εύκολα αυτά που ήδη ανέφερε ο Πέτερ Λίσε Συμφωνώ με όλα όσα είπε. Δεν θα το κάνω λοιπόν αυτό. Θα εστιαστώ επί ενός στοιχείου του σχεδίου συμφωνίας ΙΚΑΟ. Στο μέσο της αγοράς και τι κρύβεται πίσω από αυτό. Πολλά βασίζονται στην εξισορρόπηση των συνεπειών και έχουμε κάποια εμπειρία αυτής της προσπάθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εξισορρόπησης. Με στεναρότερη διατύπωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα δήλωνε ότι όλη αυτή η προσπάθεια εξισορρόπησης οδήγησε στην κατάρρευση της αγοράς άνθρακα στο εμπόριο εκομών άνθρακα της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το ETS. Οπότε είχαμε πάρα πολύ αρνητικό αντίκτυπο, όχι μόνο για το ETS, αλλά και στην καταπολέμηση των φαινομένων των κλιματολογικών το σύστημα CDM. Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την οικοδόμηση νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας με άνθρακα στην Κίνα ή στην Ινδία, διότι αντικαθιστούν παλιές μονάδες παραγωγής ενέργειας με βάση το άνθρακα. Χρειάζονται λιγότερο, παράγουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι παλιοί, αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλη πρόοδος. Πολύ συχνά είναι πρόβλημα παρά λύση αυτή η διστάθμιση των εκπομπών. Ερώτηση. Με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει να καθορίσει σχετικά κριτήρια για να αποφευθούν λάθη του παρελθόντος. Ίσως εγώ θα ήμουν πρόθυμος να προχωρήσω, αλλά μόνο, μόνο αν έχουμε αυστηρότατα κριτήρια για το θέμα αυτό της αντιστάθμισης των αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ. Κατερίνα Κομέτσνα για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ Προέδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Ξέρω ότι ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο και πολλοί συνάδελφοι προφανώς έχουν πολλές ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας. Είναι γεγονός ότι η αεροπορία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, αλλά κανείς δεν ήθελε να θίξει το πρόβλημα αυτό. Όπως και οι συνάδελφοι, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε έναν παγκόσμιο μηχανισμό, ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέσα και ελπίζω να μπορέσετε να διαπραγματευτείτε κάτι τέτοιο στο πλαίσιο του ΙΚΑΟ. Από την άλλη θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την εισαγωγή νέων καυσίμων στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι σαφές ότι Ε, η βιολογική κυροζήνη ήδη χρησιμοποιείται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Πιστεύω ότι και στην ευρωπαϊκή αγορά θα μπορούσαμε να κινήσουμε τη διαδικασία αυτή. Σας ρωτώ λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε για να χρησιμοποιείτε περισσότερο η βιοκυροζήνη ε, στις αερομεταφορές. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και πολλές θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι ε, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Μπορούμε επίσης να κάνουμε κάτι για να μειωθούν οι εκπομπές. Το πρόβλημα λοιπόν που βρίσκεται πολλές ε, χώρες χρησιμοποιούν βιοκυροζίνη, κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει ακόμα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πρασίνους, ο επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ Επίτροπε Μπούλτς, λέει ο κ. Σεκχάουτ, για την εισαγωγή που κάνατε. Είπατε ότι χαζόμαστε παγκόσμιες εμβελίας λύσεις. Συμφωνούμε στην αίθουσα. Αυτό είναι ο στόχος. Είπατε επίση ότι χρειάζονται συμβιβασμοί. Όλοι το κατανοούν. Είμαστε πολιτικοί. Καθημερινά αυτό κάνουμε. Βέβαια υπάρχει κάποια στιγμή που κάποιο λέει μέχρι τώρα βρίσκω συμβιβασμού. Παραπέρα τι γίνεται. Ήδη η ανάπτυξη ουδέτερη στον αφορά τον άνθρακα μετά το 2020 είναι τεράστιο συμβιβασμό που είναι πρόθυμη να δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πραγματικέ διαπραγματεύσει όμω πρέπει να ξεκινήσουν και ήδη κάνουμε τεράστιε παραχωρήσει. Γι' αυτό θα έλεγα ότι ήδη συμβιβαζόμεθα και πολύ μάλιστα. Και το άλλο αυτό για την παγκόσμια εμβέλεια λύση. Βλέποντα όμω τι κάνει ο ΙΚΑΟ και ο ΑΕΜΟ μέχρι τώρα η ταχύτητα των αλλαγών καθορίζεται στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Αυτοί οι οργανισμοί έτσι εργάζονται. Το είδαμε στον IMO την περασμένη εβδομάδα. Διεξήχθηκε συζήτηση για τη μείωση των εκπομπών, αλλά τα χάλασαν όλα και σε μετακύλησαν την επόμενη συνάντηση σε ένα εξάμεινο και δεν έκανε τίποτα. Και στη, στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών είναι έτοιμοι να κάνουν περισσότερο από ό,τι είναι έτοιμος να κάνει ο φορέας ο ΑΕΜΟ, το ίδιο και στον ΙΚΑΟ. Τι δεχόμαστε, αυτό δεν θα ξέρω. Αν δεν υπάρχουν πρότυπα για την αποδοτικότητα του διοξίδιου του άνθρακα. Ζητούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλεγε ότι αυτή η συμφωνία ήταν ορόσημο αυτή η συμφωνία, έτσι είπατε. Ορόσημο, συμφωνία ορόσημο, για ένα θέμα όπου τα πιο αναποτελεσματικά αεροσκάφη θα παράγονται μέχρι το 2028. Αυτό δεν είναι τόσο σημαντική συμφωνία. Λέτε ότι θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε 650 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακος. Μισό από αυτό γίνεται επιθελοντικής βάσος και το γνωρίζετε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δηλώσεις της ανακατεύει τους αριθμούς και θεωρεί ότι αυτή είναι μια καμπή η συμφωνία. Δεν είναι. Και δεν είναι αυτό που περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις επικείμενες για τα πρότυπα διοξείδου του άνθρακα. Λοιπόν, η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ ίσως να προχωρήσει πιο πέρα από αυτά που είχε συμφωνηθεί με την ΕΚΑΟ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει με τη ΣΥΠΑ σε αυτό. Στο σε παγκόσμιο επίπεδο συμφωνία, ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ, τι θα δεχτείτε. Πραγματικά ζητούμε και απαιτούμε οι εξαιρέσει για την ανάπτυξη του ανωδέτου μετάφρακα. Ότι θα προβλέπει εξαιρέσει για χώρε. Άρα χρειάζεται κάποια διθάθμιση από άλλου ο Πίτερ Λίζη το είπε αυτό. Θα το πολεμήσουμε, θα χαράξουμε κόκκινη γραμμή. Αυτό που έλεγε και ο κύριος Βαντεμπράντη για, το, για την αντιστάθμιση, offsetting. Δεν θέλουμε να γίνονται, να ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Και κάτι άλλο, να μην δεχόμαστε διατύπωση στην συμφωνία που θα απαγορεύει περιφερειακά μέτρα. Διότι ξέρουμε ότι κάποιοι λένε ότι δεν θέλουμε κανένα περιφερειακό μέτρο. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στραφεί κατά αυτού. Η δεμή θα έχετε προβλήματα στο Κοινοβούλιο προσπαθώντας να περάσετε ένα νέο ναι, μια νέα ναι, αναστολή μέτρων, stop the clock. Θα ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο θα πολεμήσει για αυτά τα θέματα και ελπίζω ότι θα καταστήσετε σαφείς τις δικές σας κόκκινες γραμμές, τα δικά σας όρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία για το EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε Μπούλτς. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ήθελα, εν συντομία, να αναφερθώ στα μέτρα της αγοράς. Επιδιώκουμε ε, να έχουμε εργαλεία της αγοράς για να πετύχουμε στόχους περιβαλλοντικούς σε κάποιο βαθμό να βελτιώσουμε τι συνθήκε που επικρατούν στον πλανήτη. Κατά την άποψή μου, μέχρι τώρα, είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα μηχανισμών που δεν λειτουργούσαν. Το ίδιο το ETS, κατά την άποψή μα, ένα μηχανισμό που δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δηλαδή, μείωση των εκπομπών που ελπίζαμε. Υπό το φως αυτών, συμφωνώ με αυτά που υπόθηκε μέχρι τώρα σχετικά με τα μέτρα αντισταθμίσεως είναι άλλη μια, άλλο ένα νιωστό στοιχείο που δημιουργεί ανησυχίες μεγάλες. Να αντισταθμίσουμε δεν είναι αποτελεσματικό μέτρο. Οι εκπομπές πρέπει να κοπούν, να μειωθούν. Πέρα από αυτό, έχω μια ερώτηση όσον αφορά την έννοια της τεχνολογικής ουδετερότητας. Συνεχώς προωθούμε αυτή την αρχή όταν ίσως θα έπρεπε να ευνοήσουμε τις τεχνολογίες που πραγματικά έχουν καλύτερη συνέπειες στο περιβάλλον. Αντί να τις ε, υπονομεύουμε. Τέλος. Πέρα από τη συμφωνία, την ενδεχόμενη που θα συναυθεί εντός ΙΚΑΟ, η Ευρώπη προτίθεται να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα. Πρόσθετες δράσεις για τη μείωση των εκπομπών από τις αερομεταφορές. Κοινοτική εναρμονισμένη δράση Φερρυπίν, που θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να εξαλείψει τις φορολογικές εξαιρέσεις για τα κάψιμα, για τον τομέα, που σήμερα ευνοείται από αυτό. προβλέπονται κάποια συμπληρωματικά μέτρα από πλευράς Ευρώπης πάνω σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να ζητήσουμε από την Επίτροπο να απαντήσει στις ε, ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, <clears throat> τις προκλητικές παρατηρήσεις ε, συχνά. Χαίρομαι που όλοι συμφωνούμε ότι δεν πρόκειται για εύκολες διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι κοινεί εμένα και τις υπηρεσίες μου. Είμαστε μέρος της διεθνούς κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ζει αποκλεισμένη πάνω σε τούτο το πλανήτη με τη δική της φιλοσοφία. Θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε αρκετά ισχυροί, ώστε όχι να πιέζουμε τους άλλους, αλλά να τους προσκαλούμε. Με μια σωστή πρόταση δηλαδή, να καλέσουμε τους άλλους να συμμετάσχουν, ε, να ε, συμβάλλουν στις προσπάθειές μας. Από τότε που ξεκίνησα τη θητεία μου ως Επίτροπος, ε, αυτό είναι το πνεύμα των εργασιών μου. Θέλω να βρούμε μια λύση κοινή αποδοχής τον Σεπτέμβριο στο Μοντρεάλ. Τα στοιχεία που έχουμε επιτάπητος αυτή τη στιγμή είναι θετικά. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλή η δομή. Επικεντρωνόμαστε στη διακυβέρνηση. Στους ε, καλούς κανόνες, στα αντισταθμιστικά μέτρα, τα offsets και σε αυτό το θέμα. Έχουμε ακόμα σκλήρες διαπραγματεύσεις. Ε, η αεροπορία όμως δεν είναι ο μόνος τομέας με αντισταθμιστικά μέτρα. Ε, μαθαίνουμε από άλλους τομείς. Ε, και νομίζω ότι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά τα μέτρα αυτά στην αεροπορία, στις αερομεταφορές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πως μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω στα αντισταθμιστικά μέτρα. Πάντω θετικό είναι ότι δεν άκουσα κανέναν να λέει ότι διαφωνεί. Από την άλλη, είναι θετικό ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφωνούν ότι διαπραγματευόμαστε επί της βασικής αρχής ε, και είναι θετικό το ότι επιδιώκουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού. Εγώ ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο φέτος, αλλά υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτές θα πρέπει να δεχτούμε ότι κάποιοι θα χρειαστούν μεταβατικές περιόδους και ότι θα ισχύσουν ε, εξαιρέσεις ε, για τις πολύ φτωχές χώρες με πολύ χαμηλό ΑΕΠ και επίσης για πολύ μικρές αγορές όπου θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρό, υπερβολικά δαπανηρό να εφαρμοστούν οι κανόνες που προτείνουμε. Αλλά θέλω να έχουμε μια διεθνή πλατφόρμα με αρκετά φιλόδοξα σχέδια στα οποία να μπορούν να συμμετέχουν όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτό θα αποτελέσει σημαντική επιτυχία. Και ναι, θα διαπραγματευτούμε και γι' αυτό χρειάζομαι την υποστήριξή σας. Θα πρέπει να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε να πείθουμε τους εταίρους μας ότι αυτή η λύση δεν είναι μόνο καλή για το περιβάλλον αλλά και για τις επιχειρήσεις, διότι ο οικολογικός προσανατολισμός σήμερα είναι ε, καλή δουλειά. Ε, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα, με την ε, ενεργειακή ανεξαρτησία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ναι, στηρίζουμε και τα βιοκαύσιμα. Έχω συναντηθεί με τον τομέα αυτών ε, μου είπαν τι όγκους μπορούν να παράγουν στο προβλέψιμο μέλλον ε, και δεν είναι τεράστιο ο όγκος αυτός ε, και άσχετα από το πόσο επιταχύνουμε τις διαδικασίες δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών μας. Ναι, καταβάλουμε προσπάθειες για τη συμπερίληψη των βιοκαυσίμων. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να ε, ασχοληθούν με τη στρατηγική για τα βιοκαύσιμα με βάση την ε, προσέγγιση των κρατών μελών θα αναλάβουμε περαιτέρω δράση. Πιστεύω ότι η συμφωνία για ε, το διοξίδιο του άνθρακα αποτελεί ορόσημο. Ήταν παγκόσμια συμφωνία μπορούμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε περαιτέρω και ποια είναι η πραγματική ουσία. Αλλά τον Φεβρουάριο είχαμε συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα όμως να έχουμε μια συμφωνία την οποία να μπορούν να ακολουθήσουν όλα τα κράτη. Ο ΙΚΑΟ έχει πάρα πολλά μέλη. Θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά την κατάσταση ώστε να καλύψουμε το κενό. Και γι' αυτό, όπως σας είπα και πριν, είναι... Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε τη συγκεκριμένη προσέγγιση και ότι ε, εργαζόμαστε με βάση την ε, μη διάκριση και τους καλούς περιβαλλοντικούς στόχους. Και ναι, το σύστημα εμπορία εκπομπών της Ευρωπαϊκή Ένωσης αποτελεί σημαντική επιτυχία. Υπάρχουν και άλλες χώρες στον κόσμο που ακολουθούν τι ε, θετικέ εμπειρίε μας και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με παρόμοιο τρόπο στο δικό τους πλαίσιο. Χρειαζόμαστε όμως μια παγκόσμια συμφωνία και ο ΙΚΑΟ εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση δεν ασχολείται με το εσωτερικό των διαφόρων αγορών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να καταλάβουμε όλοι ότι οτιδήποτε αφορά το εσωτερικό της αγοράς στην Ευρώπη θα πρέπει να μας απασχολήσει μετά τη σύναψη της συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο συνάδελφος Κανιέτ θα ε, προσπαθήσει να δει τι μπορεί να κάνει με βάση τα αποτελέσματα που θα φέρουμε από τη συμφωνία αυτή. Και νομίζω ότι τότε θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις για να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά με τρόπο ισορροπημένο. Όσον αφορά τα πρότυπα για το διοξείδιο του άνθρακα, μία παρατήρηση ακόμα. θα διαχειριστούμε το θέμα αυτό μέσω του ε, ρυθμιστικού περιβάλλοντος, αλλά νομίζω ότι και οι δυνάμεις της αγοράς θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Όσο έχουμε συνεχή πίεση, θα έχουμε και εξελίξεις. Και χαίρομαι που ακούω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι θα πρέπει ε, να ενσωματώσουμε στην τελική λύση την συνεχή αναθεώρηση ώστε να μπορούμε να έχουμε περαιτέρω συζητήσεις και περαιτέρω δράσεις με βάση το αποτέλεσμα. Είμαι υπέρ της προσέγγισης αυτής, είμαι υπέρ ενός συστήματος που συνεχίζει να εξελίσσεται με βάση το ε, ε, ποσοστό απορρόφησης στην κοινωνία. Και ναι, είμαι υπέρ των φιλόδοξων στόχων, αλλά θα πρέπει να είναι και ρεαλιστική. Σας παρακαλώ λοιπόν εμείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ε, δραστηριοποιηθούμε και να δούμε πόσο μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό θα ήθελα. Άλλα μέτρα όπως αναφέρατε. Αναφέρθηκα ήδη στο ΣΕΖΑΡ το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ε, το SES2+. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω στο θέμα αυτό και επίσης ε, το καλοκαίρι θα έχουμε μια ανακοίνωση για την απαλλαγή των μεταφορών από διοξίδιο του άνθρακα. Βλέπετε ότι ε, επενδύουμε όλο και περισσότερο στις τεχνολογίες που συνδέονται με την απαλλαγή της οικονομίας από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, χάρηκα πολύ με την ανακοίνωση της EasyJet ότι δοκιμάζει ένα σύστημα που να βασίζεται σε κυψέλες υδρογόνου. Επίσης ε, χαίρομαι με τις εξελίξεις γενικά που αφορούν τις κυψέλε υδρογόνου ε, στον τομέα των αερομεταφορών. η σημαντικότερη πρόκληση και το επαναλαμβάνω αυτό ε, θα είναι να έχουμε υβριδικό αεροσκάφος μέχρι το 2030. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε σημαντικές αλλαγές στις αερομεταφορές δεδομένης της ανάπτυξης οτιδήποτε άλλο θα είναι απλά υποστηρικτικές δράσεις. Θα προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας, αλλά η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Έχουμε κάποια μαγική λύση στα χέρια μας, όχι. Αλλά βλέπω να υπάρχει τόση βούληση που δεν έχω αμφιβολία ότι θα καταλήξουμε σε μία λύση, ότι θα συνεχίσουμε να προοδεύουμε και δεν θα τελειώσει ποτέ η διαδικασία αυτή, θα είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Δέχομαι την απεσιοδοξία σας, ασχολείστε πολλά χρόνια με το θέμα αυτό, μια δεκαετία είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά νομίζω ότι Βρισκόμαστε στην πιο κατάλληλη χρονική στιγμή και βασιζόμαστε στα αποτελέσματα της ε, Συμφωνίας COP21. Και άλλωστε τώρα πια είναι προφανής ε, οι συνέπεια της αλλαγής ε, του κλίματος. Φαίνονται στη Γρυλανδία, στη Φλόριντα. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να προσποιούμαστε. Άσχετα από το ποιος προκαλεί την αλλαγή του κλίματος, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες και να προσαρμοστούμε σε αυτήν. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, να δραστηριοποιηθούμε, να είμαστε αισιόδοξοι, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, να βασιστούμε στην κοινή μας βούληση και να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε και τους εταίρους μας να συμμετάσχουν στην επίτευξη των στόχων μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι μια πολύ καλά ανεπτυγμένη γεωγραφική περιοχή και θα πρέπει να φροντίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να συνεργαστούν μαζί μας όσοι δεν έχουν φτάσει ανάλογο επίπεδο, διότι δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας, αποκλεισμένοι από όλους τους άλλους, να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αλλαγής του κλίματος και της απαλλαγής της οικονομίας από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο κύκλο ερωτήσεων από τους ομιλητές. Ο Ιβο Μπέλετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Πολύ σύντομα να σας πω. Εγώ συμμετείχα ε, τον προηγούμενο μήνα στην ε, κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στο Μοντρεάλ. Να πω κάτι για τη διακυβέρνηση του ΙΚΑΟ. Μας προειδοποίησαν εκ των προτέρων Παρ' όλα αυτά μας εξέπληξε η έλλειψη διαφάνειας που κυριαρχεί σε αυτόν τον οργανισμό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας συμβολή. Μιλάμε για έναν οργανισμό του ΟΗΕ. Η διαφάνεια θα έπρεπε να είναι 100% ε, κάτι που δεν συμβαίνει. Είπατε για το Παγκόσμιο Αγορακεντρικό Μέτρο ότι αυτή τη στιγμή ε, ενδεχομένως θα ήταν ε, η καλύτερη δυνατή επιλογή που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η ETS, αλλά πάντως είναι ένα βήμα. Είπατε για τα, για τα πρότυπα διοξιδίου του άνθρακα, που επίσης δεν είναι πάρα πολύ φιλόδοξα, αλλά εν πάση περιπτώσει συνιστούν για κάποια πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Και δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σας κάνω. Πρώτον, για την ποιότητα των αντισταθμίσεων. Προφανώς είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό σε συνδυασμό με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητα των αντισταθμίσεων για την αξιοπιστία ε, του όλου συστήματος. Μπορείτε εσείς να εγγυηθείτε ότι πράγματι είναι υψηλή η ποιότητα αυτού του μηχανισμού. Γιατί εμείς ε, καταλάβαμε στο Μοντρεάλ τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει μια κοινή αντίληψη για το συγκεκριμένο θέμα μεταξύ των εταίρων. Επίσης είπατε ότι αυτή η συμφωνία θα προβλέπει την, την τακτική αναθεώρηση. Αυτό είναι επιλογή ή έχει ενσωματωθεί αυτό το στοιχείο στην συμφωνία. Γιατί συμφωνώ και εγώ με τον Πέτρε Λίζε και τον Ματίας Γκρότε ότι πολλές φορές μιλούμε για τις συμβολές των άλλων κλάδων και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους άλλους κλάδους ότι η αεροπορία δεν θα κληθεί να καταβάλει ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες. Ενδεχομένως θα έπρεπε να, ε, να ε, ε, να θεσπιστούν ακόμα μεγαλύτερες υποχρεώσεις, πιο αυστηρές υποχρεώσεις για τις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις, προκειμένου να δοθεί κάποιο περιθώριο ε, και στους άλλους κλάδους να ανταποκριθούν στις δικές τους ευθύνες. Ο κύριος Σεπτάνς. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει συμφωνία σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Και εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στις διατάξεις αντιστάθμισης και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια διαδικασία όπου δεν θα τίθενται στο επίκεντρο των προσπαθειών μόνο συγκεκριμένη κλάδη. Δεύτερο θέμα που με απασχολεί είναι η ενσωμάτωση του ETS σε ένα παγκόσμιο ευρωκεντρικό μέτρο. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει μια, ένα παγκόσμιο βάθρο πάνω στο οποίο θα, μπορούσαν, θα μπορούσε ο καθένας από την πλευρά του να λάβει επιπλέον μέτρα. Αλλά εμείς θέλουμε αυτό να είναι ένα βάθρο και όχι ένα ανώτατο όριο αυτό που στο οποίο θα καταλέξουμε. Ε, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο ζήτημα της διαφάνειας. Ο Ιβο Μπέλετ αναφέρθηκε ε, στις εμπειρίες μας ε, στην ε, διάρκεια αυτής της αντιπροσωπείας και της επίσκεψής μας. Προφανώς είναι απαραίτητο να, υπάρχ, να έχουμε εταίρους οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν. Δεν μπορεί να, να ε, επιβαρυνθεί ένας και μόνο κλάδος με την επίλυση του προβλήματος. Και ε, φαίνεται ότι ο τρέχον μηχανισμός, ο, τρόπο, ο τρέχον τρόπος με τον οποίο ε, χειριζόμαστε της την αεροπορία έχει λάβει υπόψη του τις ε, τεχνολογικές εξελίξεις. Τι θα κάνει η Κομισιόν προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία στο μέλλον θα είναι πολύ πιο διαφανής και ότι θα υπάρξει, μια, θα υπάρξει εμπειρογνωμοσύνη που θα κοινοποιηθεί και στον ΙΚΑΟ, αλλά όχι μόνο στον ΙΚΑΟ. Γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι κρίσιμο για να επιληθούν τα προβλήματα που αναφέρατε κι εσείς. Γιατί όπως είπατε, για την επίλυση των ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και, αυτό, και η, ο τρέχον τρόπος οργάνωσης του ΙΚΑΟ αποτελεί εμπόδιο σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Η Ζακλίν Φώστερ. Καλώς ορίζω την Επίτροπο των μεταφορών. Κρίμα που δεν ψάξαμε για παγκόσμια λύση εδώ και 10 χρόνια. Το είπε ο Πίτερ Λίζε. Κάποιοι από εμά περάσαμε αυτέ τι πολύ κουραστικέ συζητήσει επί σειρά ετών, επί σειρά ώρων, σε ατέρμονε συζητήσει, χωρί λογικό αποτέλεσμα. Όμω ίσω να είμαστε καθοδόν τώρα. Συναντήθηκα σήμερα το μεσημέρι με τον Τόνι Τάιλερ από την Ιάτα Κι άλλοι και εμπειρογνώμονε. Το κουβεντιάσαμε και το μέστε θέλει λύση. Διότι υπάρχει έλλειψη βεβαιότητας, υπάρχει καλή θέληση τώρα που το κουβεντιάζουμε. Έχω, ξέρετε το ιστορικό μου όσον αφορά τι αερομεταφορέ και την αεροπορία γενικά σε αερομεταφορέ. Δεν Έχουμε αλλάξει το σχεδιασμό των οσκαφών, των κινητήρων, των ανατράκτων, των τροχών. Κάναμε έρευνα για καύσιμα, για τα αεροσκάφη. Δεν λάβαμε υπόψη όλες αυτές τις αλλαγές για να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακος. Εμείς δεν κάναμε πολλά, το έκανε βιομηχανία. θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο δρομικό σε κάτι μέλη, όπως είναι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης. Ε, να βελτιώσουμε λοιπόν την ελληνική κατάσταση. Να έχουμε το Σέζαρ συν και το Σέζαρ, έχουμε τεχνολογία ε, και ανταγωνιζόμαστε τα αμερικανικά συστήματα. Δεν υπάρχει επαρκής βούληση από πλευράς κρατών μελών. Αν κινηθούμε όλοι μαζί, θα μειώσουμε τα προβλήματα που συζητήθηκαν ερχόμαστε στα λεγόμενά σας. Θα πάει αντιπροσωπεία α, του Κοινοβουλίου της Επιτροπής μας που θα μεταβεί στο ΙΚΑΟ τον Μάιο. Ελπίζουμε τελικά να καταλήξουν σε μέτρα με βάση την αγορά. Επιβεβαιώνεται ότι δεν θα υποχρεωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσουμε μέτρα που ξεπερνάν τα συμπεφωνημένα με την ΙΚΑΟ. Δεν θέλω περιφερειακές λύσεις που ξεπερνάνε τα όρια. Γι' αυτό καταλήξαμε σε προβλήματα πρώτη. και έχουμε μείνει πίσω, Γυρίσαν πίσω 10 χρόνια. Χρειάζονται εξαιρέσει όπω είπαμε. Υπάρχουν πολύ φτωχέ περιοχέ όπω στην Αφρική. Το δέχομαι. Γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι έχουμε την Κίνα και τη Ρωσία που δεν θέλουν να κινηθούν. Βγάλτε το Ιράκ έξω από, τον, από την εξίσωση. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα τον ανταγωνισμό όταν κάποιες χώρες δεν συμμορφώνονται. Θέλουμε λύση. Ίσως δεν έχετε σχόλια σε αυτή τη φάση. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις όμως. Τι γίνεται όταν δεν συμμορφώνονται τρίτες χώρες. Είναι ένα άλλο θέμα. Αυτά είναι τα γενικά σχόλια. Καλή τύχη εύχομαι. Ξέρετε ότι έχετε την υποστήριξή μας για την εξέβρεση λύσεως. Διότι θα θέλαμε να αλλάξουμε και θέμα. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέτρα να μειώσουμε τα αποτελέσματα. Πρέπει ανοιχτά να συζητήσουμε και να ενημερώσουμε σχετικά και τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Thank you very much, Miss Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ας ε, ω πολιτικό που ασχολείται περισσότερο με το περιβάλλον ε, και ως τέτοια δεν περιμένω να ακούσω τίποτα άλλο από αυτά που είπατε, διότι όταν θέλουμε ε, διεθνείς συμφωνίες ε, δεν μπορούν να είναι τόσο φιλόδοξες όσο ότι μπορούμε να πετύχουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύρια Επίτροπε, είπατε αποτελεί βήμα προόδου στο COP21 στο Παρίσι συμφωνήσαμε και τώρα κάνουμε ένα περαιτέρω βήμα για κοινή κατανόηση. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να πείσει έναν πολιτικό που ασχολείται ιδιαίτερα με το περιβάλλον. Ε, για παράδειγμα, ε, όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας ε, κατά το πολύ 2%, εγώ θα ήθελα ε, η, αύξηση, η μέγιστη αύξηση να ανέρθει στο 1,5% διότι αλλιώς ούτως ή άλλως θα χαθούν νησιά και θα είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή. δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον υπόλοιπο κόσμο. Μάλιστα είχαμε μποϊκοτάζ ε, με την ε, διακήρυξη της ε, Μόσχας. Γι' αυτό συμφωνώ μαζί σας ότι ναι, φυσικά είναι πάντα καλύτερο να πετύχουμε τη συμμετοχή όλων των άλλων. θα πρέπει όμως να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αποτελέσουμε εμείς στην Ευρώπη καλό παράδειγμα για τους άλλους για να τους κινητοποιήσουμε για περαιτέρω αποτελέσματα. Επίσης, ε, όσον αφορά ε, τον ΙΚΑΟ και ε, την ανάπτυξη με οδέτερο ισοζύγιο άνθρακα που θέλουμε να έχουμε μέχρι το 2020. Αυτό με τι σχετίζεται με άλλα καύσιμα, με πελτιστοποίηση των διαδρομών, μείωση των εκπομπών στα ίδια τα αεροδρόμια. Είναι δυνατόν να γίνουν πολλά, όχι μόνο όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ε, και όπως άλλωστε είπε και η κυρία Φώστερ μπορούμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα ε, σε πολλά θέματα. Σε τι βαθμό γίνονται ανταλλαγές απόψεων και για όλους αυτούς τους τομείς στο πλαίσιο της ΙΚΑΟ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλον που να θέλει το λόγο. Επίτροπε, έχετε το λόγο για απαντήσεις. Thank you very much again for... Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις. Επανειλημμένα τέθη ένα θέμα. Η διαφάνεια. Συμφωνώ 100%. Για τα πάντα. Διαφάνεια για τα πάντα. Αυτή είναι και η απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 100% διαφάνεια. Για να μπορέσουμε να εργαστούμε κιόλα. Και θα καλέσω την ΙΚΑΟ να ακολουθήσει το παράδειγμα αυτό. Η διαφάνεια και η είναι σημαντικό κομμάτι του πακέτου αυτού. Γιατί το χρειαζόμαστε. Και ελπίζω να μην υπάρξουν δυσκολίες. Διότι τα κράτη-μέλη είναι ο εφαρμοστικός φορέας. Αν δεν υπάρχει έλεγχος έχουμε πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη. Ποιο ζητάει τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση. Ποιο τα ζητάει. Για να ξέρουν ποιο ζητάει τι. Το ξέρουμε, το φροντίζουμε. Δεν νομίζω να υπάρχουν αμφιβολίες από αυτού. Όλοι επιθυμούμε, διαφάνεια στη διακυβέρνηση και στη διαχείριση. Θέλουμε σωστή εφαρμογή και υλοποίηση. Η ποιότητα της αντισταθμίσεως είναι ένα καλό παράδειγμα για διαχείριση και διαφάνεια. Πρώτο κριτήριο ποιο είναι, ότι η αντιστάθμιση θα πρέπει να είναι νόμιμη. Να μην γίνεται διπλός υπολογισμός και διπλές αξιώσεις να μην υπάρχουν. Το διαπραγματευόμαστε. Κινούμεθα όμως σωστά, προς σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω να συμμετάσχετε κι εσείς, να μας στηρίξετε διότι μετράει η φωνή σας και θα μετρήσει. Πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες του ΙΚΑΟ και θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε και τον ΙΚΑΟ να ε, στηρίζει τη διαφάνεια. Είναι φορέα του ΙΕ και δεν θα πρέπει να είναι δύσκολο. Ταυτόχρονα, εφόσον διαπραγματευόμεθα, θέτουμε επανειλημμένα το ζήτημα για να γίνει κατανοητό ότι είναι σημαντικό. Σας καλούμε και εσείς όταν πάτε να συνομιλήσετε με τους ομολόγους σας στο Μοντρεάλ να το εκφράσετε αυτό το θέμα, να το στηρίξετε. Δεν υπήρξαν πολλές ερωτήσεις, πραγματικές ερωτήσεις. Ετέθηκε το ερώτημα των ε, διαφορετικών τεχνολογιών και τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με τον ΙΚΑΟ. Μιλάμε για τα βασικά στοιχεία, για, τους, για τα δρομολόγια, ε, για τις διαδρομές, για τους μεταφορείς και σωστό επιμερισμό των βαρών και εφόσον δεν έχουμε συμφωνήσει απόλυτα, ε, δύσκολο να κάνουμε εικασίες για τα τελικά αποτελέσματα. Ίσως το επόμενο βήμα, όπως είπατε, επόμενο βήμα θα είναι τα αεροδρόμια. Καλή ιδέα είναι αυτή. Μπορούμε να το διερευνήσουμε στο μέλλον. Όπως είπα, θέλω να παραμείνω πραγματιστική στη θεώρησή μου. Έφυγε ο συνάδελφος που θέσε το θέμα. Πιέζουν οι πράσινοι, άρα θα έχουμε και μεγάλες φιλοδοξίες υπ' αυτή την πίεση. Ας μην αμφιβάλλουμε, ας έχουμε πάντα υπόψη το στόχο. Μία συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αναγκαία. Είναι ένα εργαλείο για περαιτέρω ανάπτυξη των φιλόδοξων στόχων μας. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος και να μειώσουμε την χρήση και εκπομπή του άνθρακα. Η τεχνολογία κινείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Καλύτερα υλικά, καλύτερη διαχείριση, καλύτερο σχεδιασμό. Κινείται. Η βιομηχανία προωθεί καινοτόμα προϊόντα, χρηματοδοτεί την έρευνα και την καινοτομία και τα καταφέρνουν. Αν μπορούμε να κινητοποιήσουμε και τους πελάτες θα πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ μπορείτε να μας βοηθήσετε. Εάν γίνει αυτό, θα κινηθούμε πιο γρήγορα. Στο κάτω-κάτω πελάτης πληρώνει. Και είναι οι μόνοι που έχουν χρήματα. Όλοι οι άλλοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Έχουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να συμμετάσχουν, να συνεργαστούν μαζί μας. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα εδώ να σταματήσω. Αν μου επιτρέπετε, θα σας ευχαριστήσω. Οι κριτικές που ακούστηκαν ήταν πολύ επικοδομητικές. Είναι θετική η προσέγγιση όμως, χρειαζόμαστε θετική ενέργεια. Ας κινηθούμε ως ένας. Αν δεν συμφωνείτε κάτι που υποστηρίζουμε, να το στο γραφείο μου, να με δείτε. Τους συναδέλφους, να ξεκαθαρίσουμε τα προβλήματα αν υπάρχουν. Από τη στιγμή που θα φύγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να πολεμήσουμε όσο μπορούμε και να διαπραγματευτούμε για την καλύτερη δυνατή συμφωνία του Σεπτέμβριου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς, λέει ο Πρόεδρος, για την εδώ παρουσία σας σήμερα, για τα χρήσιμα σχόλιά σας και για τη δυνατότητα που μας δώσατε να σας υποβάλουμε ερωτήσεις και να ακούσουμε ακριβείς απαντήσεις. Θα ολοκληρωθεί η συνεδρίασή μας, επόμενη συνεδρίαση, 23 και 24 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.